μάλλον να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 4 του κανονισμού και γι' αυτό μια τέτοια αλλαγή η οποία προτάθηκε θεωρείται δεκτή.